Innanzitutto Καταρχάς να καλωσορίσουμε τον κύριο Φίγκελ που είναι ειδικό απεσταλμένος για την προώθηση της ανεξιθρησκείας ε, στην, ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 24 Ιουνίου του 2013 το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση και την προστασία της ε, αναξιδρυσκείας. Το Ευρωκοινοβούλιο ανέκαθεν στήριζε τις θρησκευτικέ μειονότητες και μάλιστα εγκρίναμε ένα ψήφισμα στις 4 Φεβρουαρίου του 2016 εντός του οποίου μιλάμε για την εξόντωση θρησκευτικών μειονοτήτων από το ΙΣΙΣ και ταυτόχρονα ζητήσαμε την, ε, ε, δημιουργία της θέσης του ειδικού απεσταλμένου για την προώθηση της ανεξιθρησκείας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 6 Μαΐου 2016 ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, διόρισε τον κύριο Φίγκελ και του ανέθεσε αυτή την ευθύνη του ειδικού απεσταλμένου για την προώθηση της ε, ε, ανεξιθρησκείας ε, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθούμε την κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μειονότητες, τις θρησκευτικέ και υιοθετήσαμε μια σειρά από ψηφίσματα που καταδικάζουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα. Σας ευχαριστούμε και πάλι λοιπόν για την παρουσία σας εδώ κύριε Φίγκελ και σε σχέση με αυτή την εντολή που έχετε λάβει και τις επισκέψεις που κάνατε στο Ιράκ, και στο Σουδάν αλλά και την Αίγυπτο και την Νοτιοανατολική Ασία. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την κατάσταση προόδου, τι συναντήσατε εκεί και τι σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον. Θα σας δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς καταρχάς να καλησπερίσω όλους σας. Είμαι ευτυχής που είμαι σήμερα εδώ. Δεν θέλω να σπαταλήσω το χρόνο σας, ε, αλλά θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη, ε, την ευγνωμοσύνη μου. Ε, φυσικά γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η εξειδρισκεία. Είναι βέβαια σχετικά σύντομο το χρονικό διάστημα αυτής της εντολής και θα εστιάσω περισσότερο στο Σουδάν και το Ιράκ. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελήφθη πέρυσι, αφού το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία ένα ψήφισμα για τις μαζικές φαγές κατά χριστιανών Ιαζίδη και άλλων εθνοτικών θρησκευτικών μειονοτήτων στη ε, εδάφη όπου ε, κατέχει το ΙΣΙΣ. Ο όρος γενοκτονία δεν χρησιμοποιείται καθημερινά δεν είναι ένα συνηθισμένο όρο, αλλά είναι πραγματικό και ιδιαίτερο γιατί αυτό που συμβαίνει σε αυτά τα εδάφη αποτελούν γενοκτονία όχι μόνο κατά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και σύμφωνα με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου του Ευρώπη, ε, του Κογκρέσου των ΗΠΑ, του Βρετανικού Κοινοβουλίου, του Αυστραλιανού Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα από ό,τι απλά να παραθέτουμε ή να καταθέτουμε τέτοιες θέσεις. Και είμαι εδώ για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί η ανεξιθρησκεία είναι ε, ένας από τους καλύτερους μηχανισμούς ε, πρόληψης ε, τέτοιων γενοκτονιών. Ο τελευταίος αιώνας είναι γεμάτος από τέτοια παραδείγματα και δεν ήμασταν αρκετά ε, αποδοτικοί στην πρόληψη ούτε στην προστασία των θυμάτων και δυστυχώς ήμασταν αδύναμοι και στην τιμωρία των εγκληματιών, των δραστών. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική, να έχουμε εκπροσώπηση και να έχουμε και μέσα για να μπορούμε να προστατεύσουμε και είμαι ευτυχή που τώρα έχουμε κατευθυντήριε γραμμές στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερική δράση την ΕΙΕΔ ότι έχουμε μια, ένα intergroup ήδη σήμερα στο Κοινοβούλιο εκδόθηκε μια νέα έκθεση για την ανεξιθρησκεία στον κόσμο. Ε, τα κράτη-μέλη επίσης κάνουν πολλά σε διεθνές επίπεδες. Εδώ υπάρχουν διεθνείς ομάδες επαφών με διπλωμάτες που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα και φυσικά υπάρχουν και ευρύτερες διεθνείς πλατφόρμες και θεσμοί όπου το θέμα είναι αποδεκτό και θεωρείται πολύ σημαντικό. Πώς και τι να κάνουμε λοιπόν. Βεβαίως η ανεξαρτησίες στον κόσμο δυστυχώς σήμερα είναι κάτι το οποίο χαίρει η μειονότηση του παγκοσμίου πληθυσμού. Σύμφωνα με διάφορες ε, συγκρίσεις μπορούμε να πούμε ε, ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική και ότι η τάση είναι αρνητική. Πολλές χώρες περιορίζουν την ε, ελευθερία πεποίθησης ή θρησκείας με πολλούς